Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξη είναι η δήλωση του Συμβουλίου για την νομική βάση του μηχανισμού αξιολόγησης της Συμφωνίας του Σέγγεν. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία οφθαλμοσύλληψης catch the eye κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Äh, Κύριε Φερχόφστατ, μπορείτε να ηρεμήσετε. Ε, μπορείτε να κάνετε μετά τις ε, έντονες ε, δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μπότσκοφ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζω την κυρία Μάλμστρομ επίσης. Έχουμε συμφωνήσει ότι η κυρία Μάλμστρομ θα λάβει το λόγο μετά από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων για τη δική της δήλωση. Οπότε το λόγο έχει η Προεδρία του Συμβουλίου με τον κύριο Μπότσκοφ. Σας δίνω το λόγο κύριε Μπότσκοφ. for Europaparlamentet, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να πάρουμε το λόγο με αφορμή τη συζήτηση αυτού του ιδιαίτερου σημαντικού θέματος. Er er Είμαστε λοιπόν σύμφωνοι καταρχάς με την απόφαση αυτή. Εμείς έχουμε έρθει στην πολιτική για να παίρνουμε αποφάσεις υπέρ των λαών μας, ακόμα και αν οι αποφάσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα θα έλεγα φιλολαϊκές. Αυτό νομίζω ότι ισχύει για το σύνολο των πολιτικών που έχουν εκλεγεί εδώ υποθέτω. Η τροποποίηση της ε, λειτουργίας της νομικής βάσης είναι κάτι, του Σέγγεν εννοώ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, το αναγνωρίζω. Είναι όμως απαραίτητο εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε απτά αποτελέσματα, τα οποία επιθυμούν οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες και πιστεύουμε ότι είναι κάτι συμβατό με τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλώ, Πρόεδρε, συνεχίστε. Υπό το φως, λοιπόν, των θέσεων των κρατών μελών, η αδίποτε άλλη θέση δεν θα μπορούσε να ληφθεί στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχει για να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες και η δημιουργία μιας κοινότητας χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες της ευρωπαϊκής ιστορίας και γι' αυτό έχουμε την ευθύνη για την ε, διατήρηση αυτού του κεκτημένου, αυτής της νίκης, να έχουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα και αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις τις οποίες έχουν πάρει. Υπάρχει λοιπόν πολιτική στήριξη για την ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης του Σέγγεν. Εδώ και ένα έτος περίπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ενίσχυση του μηχανισμού έτσι ώστε να υπάρχει θα έλεγα έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει έτσι ώστε να καλύπτουμε έκτακτες ανάγκες όπου τίθεται σε κίνδυνο η συνεργασία στα πλαίσια της Συμφωνίας Σέγγεν. Αυτό είναι το λεγόμενο πακέτο διακυβέρνησης του Σέγγεν που κατετέθη τον Σεπτέμβριο του 2011 η Πολωνική Προεδρία και στη συνέχεια η Προεδρία της χώρας μου δούλεψαν έντονα σε σχέση με αυτές τις προτάσεις, τις δύο αυτές προτάσεις στο Συμβούλιο και γι' αυτό το λόγο εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ομόφωνα το Συμβούλιο Ομόφωνα λοιπόν συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει το Σέγγεν σήμερα Συγκεντρώσαμε την προσοχή μας σε ένα κυρίως θέμα, την τροποποίηση δηλαδή της νομικής βάσεως για το σύστημα αξιολόγησης της Συμφωνίας Σέγγεν. Το 77 2 ε. Φύγαμε από το άρθρο αυτό και πήγαμε στο 70 σαν νομική βάση για τη λειτουργία της Συμφωνίας του Σέγγεν. Το Συμβούλιο πήρε την απόφαση αυτή επί τη βάση διαφόρων στοιχείων. Καταρχάς, πολιτική συμφωνία για τον μηχανισμό αξιολόγησης και η τροποποίηση, όπως είπα, για το πέρασμα από το 77-2.1 προς το 70. Θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19.7 H αγγλικό του Συμβουλίου έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι έχει υπάρξει ε, αντίληψη των θέσεων του Κοινοβουλίου από πλευράς του Συμβουλίου πριν ε, γίνει δεκτό το τελικό κείμενο. Και το τρίτο στοιχείο, η τρίτη συνιστόσα της συγκεκριμένης απόφασης είναι ότι η εισαγωγή αυτή της δυνατότητας ε, ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα θα τεθεί υποσυζήτηση στα πλαίσια του επομένου τριμερούς διαλόγου. Νομίζω λοιπόν ότι οι τροποιήσεις αυτές, του, το πέρασμα από το 77 στο 70 είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα σας πω γιατί. Καταρχάς θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αν θα έπρεπε να έχουμε πράγματι έναν ενισχυμένο μηχανισμό αξιολόγησης θα ήταν απαραίτητο να αλλάξουμε τη νομική βάση. Η άλλη δυνατότητα είναι ότι δεν θα έχουμε ένα νέο μηχανισμό αξιολόγησης πολύ απλά. Κάτι τέτοιο αποκλείεται στο Συμβούλιο. Και δεν υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη ε, επί τη βάση αποφάσεων που θα βασίζονταν αποκλειστικά στο 77. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι σαν εκλεγμένος πολιτικός και εγώ και εσείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους εκλογείς μας συγκεντρώνοντας την προσοχή μας στις ανηλυμένες μας υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές λέγουν πρέπει να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στο Συμβούλιο δεν υπήρχε παρά μόνο ένας δρόμος για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Ο δρόμος αυτός δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί. Στη συνέχεια λοιπόν της αποφάσεως αυτής θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο Υπουργών συμφώνησε για την τροποποίηση της νομικής βάσεως και εδώ θα ήθελα να εξηγήσω ότι το Συμβούλιο με την απόφαση του αυτή στην ουσία έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση επί τη βάση της γνωμοδοτήσεως της νομικής υπηρεσίας για την ουσία της υπόθεσης αυτής. Τρίτον, το Συμβούλιο διευκρίνησε με ξεκάθαρο τρόπο ότι λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που άπτονται της μελλοντική συζητήσεως της συγκεκριμένη απόφασης που μόλις έλαβε. Ελπίζω να καταλάβετε ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης της νομικής βάσεως εδράζεται αποκλειστικά σε θέματα ουσίας και περιεχομένου και όχι σε θέματα πολιτικής. Αγαπητά μέλη, του Κοινοβουλίου. Θα ήταν εντελώς λάθος να μετατρέψετε το θέμα αυτό σε σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν θα υπήρχε χειρότερο λάθος και θα ήταν κάτι το οποίο θα έβλαπτε συνολικά τη συνεργασία μας στα πλαίσια του Σέγγεν η οποία θα πρέπει να παραμείνει ισχυροτάτη. Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορέσει να συνεχίσει τον διάλογο στο σύνολο του πακέτου Σέγγεν και όχι μόνο τον έλεγχο στα σύνορα, αλλά και την πρόταση για τον μηχανισμό αξιολόγησης γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει αυτή την εποχή τρομερές προκλήσεις. Απαιτείται λοιπόν μια στενή συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Μόνο από κοινού θα δοθούν απαντήσεις και μόνο χάρη συνεργασία θα υπάρξουν λύσεις, λύσεις στις οποίες προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Προεδρία της Δανίας αποδίδει μια τεράστια σημασία στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξ αρχής είχαμε πάρα πολύ στενές επαφές με τους εισηγητές για τον μηχανισμό αξιολόγησης και με τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ακούσαμε προσεκτικά. Υποσχεθήκαμε ότι θα σας ακούσουμε και θα λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις σας. Υποσχεθήκαμε έναν διάλογο παραγωγικό και γνήσιο και πράγματι νομίζω ότι στις 31 Μαΐου η Επιτροπή Λίμπε αναγνώρισε ότι η Προεδρία έκανε προσπάθειες για να εμπλέξει το Κοινοβούλιο στις συζητήσεις, στις συζητήσεις που οδήγησαν στην συγκεκριμένη συμφωνία στο Συμβούλιο. Η πρόταση αυτή λοιπόν είναι μια πρόταση προς την σωστή κατεύθυνση κάναμε ένα βήμα προόδου και αυτό οφείλεται και στη συμμετοχή και την προσπάθεια του κυρίου Κοέλιο και των υπολείπων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί η συμβιβαστική πρόταση στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη και το σημείο της απουσίας ελέγχων σε επίπεδο εσωτερικών συνόρων ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίδεται η δυνατότητα για περαιτέρω απρόβλεπτες ε, και μη ανακοινωθήσει εκ των προτέρων επισκέψεις επιτόπου των ελεγκτικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια έτσι ώστε να ενημερώνεται με σωστό και τακτικό τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επαφές ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα είναι ιδιαίτερο στενές. Δεν εκπλήσεται κανείς λοιπόν που τα θέματα που είναι σημαντικά για την Προεδρία είναι σημαντικά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχετικά τώρα με τον κώδικα Schengen, τον λεγόμενο συνοριακό ή μεθοριακό, υπόκειται πάντα στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή τίνας συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το υπογραμμίζω αυτό, γιατί το θέμα αυτό του ελέγχου σε επίπεδο εσωτερικών συνόρων είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερο στο Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό ακριβώς η Προεδρία θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε οι πολιτικά ευαίσθητες αυτές τις αποφάσεις για τον έλεγχο ή την εισαγωγή του ελέγχου σε επίπεδο εσωτερικών συνόρων να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί πριν από το σύνολο του κώδικα Σέγγεν. Τροποποιώντας λοιπόν την κατάσταση παραμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον συνομοθέτης σε τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Ακόμα και αν η πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την αλλαγή της νομικής βάσης είναι πλέον δεδομένη. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και μία πρόταση για την μετακίνηση των ρητρών για την επανασαγωγή των ελέγχων Ε, στον μηχανισμό αξιολόγησης. Η Προεδρία εδώ δεν είχε συμφωνήσει. Εάν υπήρχε η μετακίνηση αυτή, τότε θα ήταν αυτονόητο ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει κριτική στη θέση του Συμβουλίου. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε δεκτό τελικά από το Συμβούλιο, δεν υπήρξε μετάθεση αν θέλετε των προβλέψεων και γι' αυτό συνάδελφοι εφόσον έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα αυτό είναι καρπός προσπαθειών ε, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμων και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσετε την πρότασή μας ε, με ευρύ πνεύμα παρακαλώ. Η πρόταση του Συμβουλίου, αυτό το οποίο επιθυμεί είναι να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο το οποίο να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μοντέλο το οποίο να είναι πιο κοινοτικό στο Συμβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα διαπιστώσαμε ότι αυτό το οποίο έχει σημασία για το Συμβούλιο είναι να συμμετέχει ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Σέγγεν και στην στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. Ελπίζω η συζήτηση που θα ακολουθήσει να είναι πλούσια. Όλοι όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το Συμβούλιο αυτό το οποίο επιθυμεί είναι ένα στενός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν γύρω από αυτή τη θεματολογία, μια θεματολογία καθοριστική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εμάς ανήκει συνάδελφοι και σε εννοώ και στους δύο να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η πρόταση αυτή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση με τις παρεμβάσεις των αρχηγών των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν ο πρόεδρος του ΕΛΚΟ, Ζωζεφτόλ. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν μου λείπει βέβαια η τάση να εκραγώ. Είναι μια πρόκληση κύριε Υπουργέ και κάνετε και μια πρόσθετη πρόκληση σήμερα το πρωί. Εγώ κρατάω την ψυχραιμία μου παρόλα αυτά. Με, το, με την απόφαση του Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση, αντίθετα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν το Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε να αλλάξει το μηχανισμό Αξιολόγηση του Σέγγεν, την ε, νομική του βάση συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Εσωτερικών έχουν πάρει μια απόφαση η οποία είναι απολύτω απαράδεκτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάλστρομ, η οποία δεν υπέκυψε στις πιέσει του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε, κυρία Μάλστρομ, την Κομισιόν και στη συνέχεια, γιατί θα είναι δύσκολε συζητήσει. Αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν εφαρμόσατε και ένα καθεστώς για τις προξενικές θεωρήσεις. Θα είχατε προστατεύσει έτσι καλύτερα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρωτοβουλία αυτή. Έχετε διασπάσει, έχετε διαρρήξει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε θίξει με επικίνδυνο τρόπο την βασική αρχή της κοινοτική μεθόδου. Και ξέρετε ότι εγώ είμαι προσιλωμένος ιδιαίτερα σε αυτή τη μέθοδο. Όταν επιτίθεστε εναντίον αυτή τη αρχή, θα μα βρείτε αντιμέτωπου με εσά. Η αρχή αυτή σημαίνει ότι τα μεγάλα κράτη δεν, δεν επιβάλλουν τη θέλησή τους στα μικρά κράτη και το ενωσιακό συμφέρον υπερτερεί του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό το καταργήσετε με την απόφασή σας. Η αρχή αυτή λοιπόν της κοινοτική μεθόδου είναι μια αρχή την οποία υπερασπίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν και δεν θα απαρνηθεί αυτή την στάση του. Θα ζήτησα από την κυρία Τόνινγκ Σμιτ, την πρώτη του Συμβουλίου, η οποία ήταν και ευρωβουλευτή στο παρελθόν, να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου για να εξφράσει την άποψή τη. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή σήμερα να ήταν εδώ παρούσα, γιατί είναι σημαντική η ενωσιακή μέθοδο και ξέρει η κυρία Τόνινγκ Σμιτ περί τίνο πρόκειται. Η Ιδανική Προεδρία δεν σέβεται επαρκώ τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων, ώστε να κάνει τον κόπο να πει γιατί δεν θέλει να δώσει στους βουλευτές το δικαίωμα στην απόφαση σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για, από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι από την προηγούμενη Πέμπτη έχει λήξει ουσιαστικά η Δανική Προεδρία. Εμείς θα αναφερόμαστε μονάχα στην επόμενη Προεδρία, την Προεδρία της Κύπρου. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο Χρειάστηκαν πολλέ συζητήσει και δύσκολες αποφάσεις. Αλλά εσείς έχετε παραβιάσει την κοινωνική μέθοδο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμά. Σε μια χρονική στιγμή όπου η οικονομική και η κοινωνική κρίση που διατρέχουμε ζητάει από όλους μας και από όλους τους ηγέτες Ευρωπαίους ή εθνικούς ηγέτες να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης και σεβασμού, εσείς έχετε καταστρέψει αυτό το σεβασμό με το να αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας προς το Κοινοβούλιο, πηγαίνετε σε μια κατεύθυνση που είναι αντίθετη από αυτή που θα μας βοηθούσε να βγούμε από την κρίση, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Η επίλυση των, των προβλημάτων δεν είναι να κλείσουμε τα σύνορα. Αντίθετα, είναι να έχουμε την επιμερισμένη κυριαρχία, να έχουμε ένα πνεύμα αμοιβαία κατανόησης και εμπιστοσύνης, ώστε να διασφαλίσουμε αυτά που είναι τα πιο σημαντικά για μας, τις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν ανατρέψει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο αυτή την απόφασή του, θα έχει πάντα αντιμέτωπό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Χάνες Βόμποντα, ο επικεφαλής της ομάδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ορισμένοι θα δυσκολευτούν να αντιπαρατεθούν με μια ε, σοσιαλιστική προεδρία. Αλλά μας διευκολύνεται το έργο μας. Είπατε ότι αποφασίσατε ομόφωνα όμως και εμείς απορρίπτουμε αυτήν την απόφαση. Η ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών ομόφωνα θεωρεί ότι κάνατε λάθος και ακολουθείτε επικίνδυνη πορεία από την προηγούμενη κυβέρνηση στη Δανία δεν μάθατε τίποτε, ε, δεν αντλήσατε διδάγματα ε, και από την εμπειρία σας ε, με τους δεξιούς λαϊκιστές. Δυστυχώς δεν μάθατε τίποτε και επανέρχεστε τώρα. Ε, θεωρήσατε ότι υπήρχε τεράστιο κύμα από την Τινησία. Οι ο Ιμπερλουσκόνη, οι Σαρκοζή είχαν συμφωνήσει να κλείσουν τα σύνορα. Λες και αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Πού είναι τα εκατομμύρια των μεταναστών στην Ευρώπη ε, για να αντιδράσετε. Χρειάζεται μια σωστή παρέμβαση τα εκατομμύρια μετανάστες πήγαν από τη Λιβύη στην Τινησία και πολλοί Λίβοι ε, ε, ε, επειδή πήγαν στην Τινησία πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα. Είναι δηλαδή αυτή η απάντησή μας στην Αραβική Άνοιξη. Αυτή είναι 100% λάθος αντίδραση από εμάς. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στα σύνορα. Γι' αυτό πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα. Αλλιώς δηλαδή δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν μπορούμε πια στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κάποιο στην Ευρώπη που θα μιλήσει για αλληλεγγύη, θα μιλήσει για εξασφάλιση και θωράκιση των συνόρων απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Τώρα ε, έχουμε συνηθίσει να αντιδρούμε σε λαϊκιστικά ε, αιτήματα και ε, αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να το κάνει η Δανική Προεδρία. Και πραγματικά ε, έρχεστε εδώ και λέτε ότι πρέπει να νιώθουμε και ευγνωμοσύνη επειδή μας γλιτώσατε από τα χειρότερα. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη σας για το Κοινοβούλιο. Να γονατίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε γονατιστή γιατί διαφυλάσσετε τα σύνορα. Ε, γιατί ε, ε, χρειάστηκαν οι αλλαγές και εδώ συμφωνώ με την Επίτροπο. Πάντοτε η ελευθερία την ε, διακίνηση και τόσο, τόσο συχνά την προασπίσαμε, ε, έπρεπε να σας δείξει ότι θα υπήρχε αντίδραση από εμάς αν χωρίς λόγο ξανακλίνατε τα σύνορα. Και γι' αυτό ε, θα έπρεπε να εισακουστεί το Κοινοβούλιο. Αν θυμάστε ε, τις προηγούμενες εξελίξεις θα καταλάβετε που φυσάει ο άνεμος. Κάποιοι υπουργοί θέλουν να αυξήσουν τις δυνατότητες που έχουν και στη Δανία και αλλού θέλουν να έχουν αυξημένες δυνατότητες να κλείνουν τα σύνορα. Αυτό κρύβεται από πίσω και αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Ε, και η ομάδα μας και οι άλλες ομάδες ομοφωνούν και με κάθε μέσο πολιτικό και νομικό θα αντιταχθούμε σε αυτό που κάνετε. Ανοίγετε την πόρτα για το δεξιό λαϊκισμό στην Ευρώπη και λυπάμαι πάρα πολύ που βρέθηκε να είναι ιδανική προεδρία ιστορία εκείνη που άνοιξε τη διάπλατα την πόρτα στο λαϊκισμό. Για την ομάδα των φιλελευθέρων, ο κύριος Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, την, ε, πέμπτη, την επόμενη πέμπτη, ε, εορτάζομαι την 27η επέτειο του Σέγγεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο που μας κάνατε, κύριε Υπουργέ. Παρέμβαση εκτός μικροφών. Νομίζω ότι είναι ντροπή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Είναι έσχος Έσχος κύριε Υπουργέ, όταν λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συζήτησης αυτής ε, δημοσιεύεται ανακοινωθέν στον τύπο στα δανεικά που λέει ότι η συμφωνία είναι καλή για την Ευρώπη και αποτέλεσε το αποτέλεσμα ε, σε βάθος διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό λέει η δήλωση που έγινε σήμερα το πρωί, πριν από λίγα λεπτά. Εξεδόθη από τις υπηρεσίες σας. Υπουργέ, δεν ζούμε πια στο Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα έτσι γινόταν ο διάλογος μεταξύ του βασιλιά και του των κοινοβουλίων τότε. Τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν έχουμε διάλογο. Μιλάμε για συναπόφαση στις σύγχρονες κοινωνίες και στα σύγχρονα κοινοβούλια. Δεν χρειαζόμαστε το διάλογο σας λοιπόν. Εμείς θέλουμε να αναγνωρίσετε τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται για αντιπαράθεση σε σχέση με τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι θέμα απόπειρα από το Συμβούλιο επανεθνικοποίησης του Σέγγεν, κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, αλλάζει τη νομική βάση, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρεθεί έξω από τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων και δεύτερον και πιο σημαντικό, δηλώνοντας ρητά ότι η υλοποίηση του νέου κεκτημένου θα πρέπει να ανατεθεί στο Συμβούλιο και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε δεν είναι ε, επίθεση κατά του Κοινοβουλίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινοτικής Μεθόδου και του γεγονότος ότι το Σέγγεν αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και το μεγαλύτερο σκάνδαλο ακόμα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, συνάδελφοι, που δεν είναι ε, πλήρως στο Σέγγεν, που έχει επιλέξει να είναι εκτός, θα αντιμετωπίζεται καλύτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι με το άρθρο 70 θα συνεχίζουν να έχουν παρουσία στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουν λόγο από ό,τι φαίνεται, αλλά θα είναι παρόντες. Το, κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι όμως. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβουμε ξεκάθαρη δράση σήμερα. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Δεύτερον, Γιατί θα πρέπει να πληρώσουμε για όλα αυτά, αν θέλουν να επανεθνικοποιήσουν, να επανεθνικοποιήσουν και να πληρώνουν οι ίδιοι το ε, κεκτημένο του Σέγγεν και να μην το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Τρίτον, γιατί να συνεχίσουμε, Υπουργέ, ε, μαζί σας ε, στο, στις ε, δικαιοσύνη και εσωτερικά, εσωτερικές υποθέσεις. Έχουμε τριμερή διάλογο τον Ιούνιο. Γιατί να συνεχίσουμε στις 19. Γιατί να συνεχίσουμε την έκθεση Δίαστε Μέρα για την ρήτρα διασφάλισης. Έχουμε δύο τριμερεί στις επόμενες δύο εβδομάδες. Γιατί να τα συνεχίσουμε όλα αυτά. Γιατί να συνεχίσουμε με την έκθεση Βέμπερ για την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα. Και γιατί να συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα με τη Δανική Προεδρία, γιατί να μην αναστείλουμε όλες τις συνομιλίες ε, στις, ε, στη δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις ε, και να περιμένουμε μέχρι να αναλάβει η επόμενη Προεδρία. Για τους πρασίνους έχει το λόγο η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η ιδανική κυβέρνηση κάνει κάτι το οποίο ξέρει ότι είναι λάθος. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε ένα αποτέλεσμα που εγώ θεωρώ ότι ήδη οι ευρωπαϊστές στην ε, δανική κυβέρνηση που θέλαν να επιτύχουν την πρόοδο στα ευρωπαϊκά θέματα γνωρίζουν ότι είναι μια λανθασμένη αντιμετώπιση. Όταν οι Σοσιαλδημοκράτες ακολουθούν την οδό των δεξιών λαϊκιστών αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά σε κανένα καλό αποτέλεσμα. Όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο, με την ουσία, έχουν λεχθεί. Εγώ απλώς θέλω να θίξω ένα σημείο που έχω ίσα ίσα ένα λεπτό να αναφέρω. Για μένα είναι σημαντικό και είναι κάτι που με εξοργίζει το ότι μια δανεική προεδρία με την οποία η δική μου πολιτική ομάδα προσπάθησε να έχει πολύ στενή συνεργασία σήμερα έρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ευρώπης. Και δεν έχει εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στα θέματα αυτά να μπορέσουμε εμείς να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας προς όφελος των πολιτών μας. Στο Κοινοβούλιο αυτό βρισκόνται πρώην αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί, πρώην υπουργοί, γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά. Σκεφτείτε γιατί εσείς πιστεύετε ως Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας την ασφάλεια των πολιτών και δεν έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε τα θέματα αυτά. Είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδη αυτά τα πράγματα. Φαίνεται πια ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ενώ είμαστε σε μια τόσο βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση, εσείς ανατρέπετε κάτι το οποίο ήταν και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περνάτε σε ένα χώρο λαϊκισμού. Καταστρέφεται μια από τις μεγάλες επιτεύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ελευθερία διακίνησης. Αυτό είναι έσχος. Σήμερα λοιπόν δεν ισχύει αυτό το οποίο είπατε στην δήλωση του Συμβουλίου ότι είναι μια θετική μέρα για την Ευρώπη. Είναι η πιο σκοτεινή και θλιβερή μέρα της δανικής σας προεδρίας. Αντίθετα. Η κυρία Μάκιντάιρ από τους συντηρητικούς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ εξεπλάγινα από την κίνηση του Συμβουλίου να αλλάξει τη νομική βάση του Σέγγεν, αλλά ειλικρινά εκπλήσωμαι ακόμη περισσότερο από τις αντιδράσεις των συναδέλφων σήμερα εδώ. Ε, πρέπει να διατηρήσουμε τώρα την υφαλιότητά μας, να σκεφτούμε ψύχρεμα. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε παιδαριωδώς. ε, ε προκλήσεις είναι μεγάλες σήμερα στην Ευρώπη και χρειάζονται καλές σχέσεις εργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα. Το πρώτο βήμα μας θα πρέπει να είναι να διερευνήσουμε τις νομικές επιπτώσεις των ε, ενεργειών του Συμβουλίου. Πρέπει να πω ότι κατανοώ τα κράτη-μέλη που ομοφόνος ε, συμφώνησαν να αλλάξουν τη νομική βάση. Ο μηχανισμός αξιολόγησης ε, συνδέεται με την πρόταση για προσωρινούς ελέγχους στα σύνορα. Και τα δύο τα ψηφίσαμε χθες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και στις δύο περιπτώσεις είδαμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ε, μιας διακυβέρνησης του Σέγγεν με έδρα της Βρυξέλλες. Και στις δύο περιπτώσεις τα κράτη-μέλη διαφώνησαν στεναρά με πολύ στέρεα επιχειρήματα. Θα θυμάστε ε, Το άρθρο 4 ε, της Συνθήκης της Ένωσης ε, προβλέπει το, ότι το θέμα αυτό της ασφάλειας είναι ευθύνη κρατών μελών. Θεωρώ ότι η διαχείριση των εθνικών συνόρων συνδέονται άμεσα με θέματα εθνικής ασφάλειας και καταλαβαίνω γιατί τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να παρετηθούν από την εξουσία τους αυτή. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με σύνομο και ε, νυφάλιο ε, τρόπο, με ψυχραιμία, χωρίς αυτές τις άσκοπες αντιδράσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Μακίντα υπάρχει ερώτηση από τον κύριο Γκέμπελς για σας. Συμφωνείτε? Λυπάμαι. Η κυρία Μακίνταρ δεν θέλει να... δεν δέχεται την ερώτησή σας. Και τώρα, εξ ονόματος της ομάδας της ε, ε Νοτικής Αριστεράς, η κυρία Κορνέλη Έρνς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, το άνοιγμα των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σημαντικότερο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως και έχει μεγάλη ελκτική δύναμη για πολλούς στον κόσμο. Παράλληλα, ως αριστερά πάντοτε επικρίναμε το γεγονός ότι ε, κλείναμε τα σύνορα προς τα έξω. Ήταν πολύ σημαντικό για μας λοιπόν να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης και τώρα ε, τον παραβιάζει το, το Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι αυτό που γιορτάζεται ως Συμβούλιο ε, είναι λάθος. Ξαναγυρίστε στις αρχές της κοινότητας. Σας καλώ να το κάνετε αυτό θέτοντας τέλος σε μια πολιτική που είναι σε τελευταία ανάλυση αντιευρωπαϊκή. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική του Συμβουλίου εν προκειμένου είναι αντιδημοκρατική διότι Θέλει να μας υποβαθμίσει ως κοινοβούλιο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς ε, έχουμε δικαίωμα συναπόφασης βάσει της συνθήκης και θέλουμε να το ασκήσουμε εν προκειμένου. Δεύτερον, η απόφαση του Συμβουλίου είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή γιατί εθνικοποιεί το Σέγγεν. Και σας ρωτώ, ρωτώ τη Δανική Προεδρία, το Συμβούλιο, Θέλετε να εισάγετε πάλι τελωνιακά σύνορα, θέλετε να ξαναγυρίσουμε στον προηγούμενο αιώνα. Τι θέλετε να ε, προβάλλετε με την απόφαση αυτή. Γελιοποιήστε και στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Τρίτον, η απόφαση του Συμβουλίου είναι βαθύτατα λαϊκιστική και προωθεί έτσι εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν την επανεθνικοποίηση και την καταστροφή της ευρωπαϊκής διάστασης. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Σας καλώ να αποσύρετε την απόφασή σας. Ξαναγίνετε Ευρωπαίοι κυρίες και κύριοι. Για τους μη εγγεγραμμένους έχει το λόγο ο κύριος Τσάλστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη Αποφάσισαν λοιπόν να αναλάβουν εκ νέου τις ευθύνες τους για να έχουν ασφαλή σύνορα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παίξει κανένα πλέον ρόλο σε σχέση με την απόφαση αυτή. Για τους φιλελεύθερους αυτό είναι μια διακήρυξη πολέμου, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν έχει κάνει τίποτα για να εμποδίσει τους παράνομους να εισέρχονται στα ευρωπαϊκά εδάφη. Συνεπώς, για να αποφύγουν τέτοια προβλήματα, τα κράτη-μέλη αποφεύγουν την ασφαλή οδό εναντίον των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν το Κοινοβούλιο λοιπόν διαφωνεί, τότε τα κράτη-μέλη παραμένουν έτσι και αλλιώς στις θέσεις τους και δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουν οι πολιτικές αποφάσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, εκεί όπου πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το Κοινοβούλιο αυτό δεν έχει λόγο ύπαρξης για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαλυθεί. Κυρία Μάλμστρομ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Πριν από ένα χρόνο υπήρχε μεγάλη αναταραχή σε σχέση με το Σέγγεν υπήρχε κάποια ανασφάλεια για το τι θα γινόταν αν υπήρχαν συνοριακά προβλήματα. Κάτω από ποιε συνθήκε θα μπορούσαν να υπάρχουν και πάλι προσωρινή συνοριακή έλεγχη. Ζητήθηκε από την Κομισιόν να κάνει προτάσει για τη βελτίωση του Σέγγεν και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι κρίσει βάσει ευρωπαϊκών μηχανισμών. Πέρσι το Σεπτέμβριο κατέθεσε τέτοιε προτάσει η Κομισιόν κάναμε μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκού χαρακτήρα μηχανισμού αξιολόγηση, ώστε να μπορεί η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη, του εμπειρογνώμου των κρατών μελών και άλλου φορεί να ανοιχνεύσουν προβλήματα εγκαίρω στα σύνορά μα, για να μπορέσουν επίση να εντοπίσουν τι μπορεί να γίνει, να προτείνουν θεραπείε, να ενεργοποιήσουν τα μέσα στη διάθεσή μα και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράση το οποίο θα ήταν υποχρεωτικό και υπό την εποπτεία τη Κομισιόν. Αυτό θα αντικαθιστούσε την ε, εποπτεία ομοτήμων κατά κάποιο τρόπο που ισχύει αυτή τη στιγμή. Θα βασιζόταν αυτό στο άρθρο 77, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε μια στεναρή δέσμευση και θα ενισχυόταν η πολιτική νομιμοποίηση αυτής της πρότασης με τη συναπόφαση. Δεν ήταν μοναχα θέμα περιεχομένου, ήταν θέμα πολιτικής φιλοδοξίας επίση. Η άλλη πρόταση ήταν για τον κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Πάλι ένα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την επανεισ επαναφορά των μηχανισμών ελέγχου στα σύνορα ω τελική καταφυγή, εάν δεν μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα σύνορά του, αλλά το Σέγγεν είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο το γνωρίζουν και το εκτιμούν οι πολίτε. Τα σύνορα δεν αφορούν μόνο του πολίτε του ίδιου, αλλά και το εμπόριο, την οικονομική ανάκαμψη και όλα αυτά. Επομένω, δεν μπορεί να υπάρξει μια μονομερή απόφαση για να οι συνοριακοί έλεγχοι. Θα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση. Εμεί ω Κομισιόν είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση του Συμβουλίου. Δεν προσθέτει τίποτα στου τωρινού κανόνε. Δημιουργεί ένα μηχανισμό που δεν υπάρχει πραγματική απόφαση ε, εφαρμογή που να μπορεί να έχει συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε καταχρήσει ή λαϊκιστικέ καταχρήσει λόγω εσωτερική πίεση. Εγώ εκτιμώ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχει λεχθεί ο τελικό λόγο για τα θέματα αυτά. Έχουμε λάβει υπόψη επίση την ψηφοφορία χθε στην Επιτροπή ΛΕΜΠΗ, ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κομισιόν μαζί σα θα αγωνιστεί για τα θέματα αυτά. Βασίζεται στη δική σα υποστήριξη για να έχουμε ένα ισχυρό Σέγγεν προ όφελο των πολιτών μα, ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, αλλά να διατηρήσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία για του πολίτε, τι επιχειρήσει, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση κτλ. ώστε να έχουμε σαφεί ευρωπαϊκού κανόνε για την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Σέγγεν. Ευχαριστώ. Και τώρα ο του Συμβουλίου, ο κύριος Μπότσκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή η οποία είναι ιδιαίτερα ζωντανή και έντονη και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να απαντήσω άμεσα σε αυτά τα οποία ρέτησαν και να σας εκφράσω τη θέση του Συμβουλίου για το μηχανισμό του Σέγκερ. Άκουσα όλες τις απόψεις των κυρίων κοινοβουλευτικών σήμερα. Ένα σημείο το οποίο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι το ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την επανεισαγωγή ελέγχων στα σύνορα που αναφέρθηκαν σε αυτή η διάφορη κοινοβουλευτική αλλά όλα αυτά περιλαμβάνονται στην φυσιολογική νομοθετική διαδικασία, στην απόφαση. Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση και το Κοινοβούλιο διατηρεί την επιρροή του για τα θέματα αυτά. Δεν ευσταθεί αυτό το οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ορισμένοι ότι έχει λάβει χώρα, ότι υπάρχει μια διελκυνστίνδα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η τροποποίηση της νομικής βάσης είναι μια απαραίτητη συνέπεια των συμφωνιών επί της ουσίας που επέτρεψαν να υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις του για το περιεχόμενο αυτής της πρότασης κατέδειξε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε μία, την απαραίτητη πλειοψηφία για μια πρόταση η οποία θα βασιζόταν στο άρθρο 77. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Συμβούλιο αναγνωρίζει και πλήρως το γεγονός ότι και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο έχουν κοινά συμφέροντα για να δημιουργηθεί ένα σύστημα Schengen το οποίο λειτουργεί σωστά και παρέχει ασφάλεια. Από την άποψη αυτή λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο για την προσήλωσή του στα θέματα αυτά και τη συμβολή του για τη συνεργασία στα θέματα του Σέγγεν. Σε πολλέ περιπτώσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε τον αποφασιστικό ρόλο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο, σε μεγάλο βαθμό, είναι πράγματι επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το σύστημα Schengen ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Ο κύριος Κουέλιου για πολλά χρόνια υπήρξε η ενσάρκωση αυτού του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να βασιστούμε και πάλι στην δέσμευση και στη συμβολή του κυρίου Κουέλιου στα θέματα αυτά. Παρά τις διαφορές απόψεων λοιπόν που έχουν εκφραστεί σήμερα, εγώ διατηρώ την εμπιστοσύνη μου, είμαι σίγουρος ότι η απόφαση η οποία θα είναι κεφαλαιώδης θα είναι αυτή που θα δημιουργήσει το καλύτερο πλαίσιο για να υπάρχει πιο αποτελεσματική διαχείριση της, της συνεργασίας μας στα πλαίσια του Σέγγεν. Το Συμβούλιο συμφώνησε την προηγούμενη Πέμπτη για μια θέση η οποία έγινε δεκτή ομόφωνη. Ομόφωνα παραμένουμε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και πολλές από τις συζητήσεις μας για τη διακυβέρνηση του χώρου του Σέγγεν έχουν ευνοηθεί από τις θετικέ επαφές που είχαμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Δανική Προεδρία θέλει να εξασφαλίσει ότι τα αιτήματα του Κοινοβουλίου θα ληφθούν υπόψη στην τελική συμφωνία στην οποία καταλήγει το Συμβούλιο. Είμαι πεπισμένο ότι η Δανική Προεδρία σε μεγάλο βαθμό έχει επιτύχει στο να συγκεράσει όλες αυτές τις απόψεις στην τελική συμβαστική λύση. Η ελπίδα μας είναι ότι η τελική απόλυξη όλων αυτών των προσπαθειών θα είναι ικανοποιητική και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο για όλα τα θέματα διακυβέρνησης του Σέγγεν. Τώρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα, το συνοριακό κώδικα, το Κοινοβουλίο θα πρέπει να διαδραματίσει τον κλασικό του ρόλο συναπόφασης για το μηχανισμό αξιολόγησης του Σέγγεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εκφέρει γνώμη για τα τελικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου. Όπως υπεγράμμισα όμως και στην αρχική μου παρέμβαση, το Συμβούλιο θέλει ένα διάλογο για το σύνολο των θεμάτων αυτών, όχι μόνο τους συνοριακούς ελέγχους, αλλά και για το μηχανισμό αξιολόγησης. Για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε σαφές ότι το Συμβούλιο σε μεγάλο βαθμό θέλει να λάβει υπόψη απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την ε, πρόταση για, την, για το χώρο του Σένιερ και εδώ είμαι πάρα πολύ σαφής. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Το Συμβούλιο θέλει και έχει την απαραίτητη θέληση να αναπτυχθεί ο στενότερος δυνατόν διάλογος με το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι το Συμβούλιο έχει τις καλύτερες προθέσεις. Εάν το Συνοβούλιο και το Κοινοβούλιο συνενώσουν τις δυνάμεις τους, μόνο τότε θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα που είναι τα απαραίτητα αποτελέσματα και είναι αυτά που προσδοκούν οι λαοί μας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια στενή συνεργασία για το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να προκύψει ένας επικοδομητικός και στενός διάλογος μαζί με το Κοινοβούλιο και αυτό ισχύει και για τις επερχόμενες προεδρίες. Εγώ γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παρουσιάσει και τις δικές του προτάσεις για τα θέματα αυτά. Εγώ θα διαβιβάσω αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να με ενώπιόν σας για να σας κάνω μια ε, παρουσίαση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Μπόσκοφ. Ε, νομίζω ότι αυτή η πρόσκληση για συνέχιση της συζήτησης είναι μονόπλευρη. Τώρα, ε, οι ομιλητές ε, στους οποίους ε, απευθύνθηκαν άμεσα έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της συζήτησης να κάνουν μια προσωπική δήλωση. Αυτό αφορά και τον εισηγητή κύριο Κοέλιο, ο οποίος αναφέρθηκε πολλές φορές με βάση το άρθρο 151. Δίνω στον κύριο Κοέλιο το λόγο αμέσως. Παρακαλώ. Η Ιδανική Προεδρία Άρχισε καλά. Άρχισε καλά με την προσέγγιση του κυρίου Μπότσκοφ το και ε, κατέληξε όμως ότι δεν εμπιστεύεται το Κοινοβούλιο και αυτό δίνει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα ε, σε σχέση με την, και με την συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να ε, υπάρχουν έλεγχοι και κατηγόρησε το Συμβούλιο που δεν ήθελε μια πραγματική αξιολόγηση του συστήματος Σέγγεν. που θα μας επέτρεπε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε ε, για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Κατηγορώ το Συμβουλίο που θέλει να ε, διατηρήσει το σύστημα, όπως ε, είπε και πολύ σωστά η Σεσίλια Μάλμστρεμ. Αποκρύπτει ή παραγνωρίζει τα λάθη και τα προβλήματα. Δεν θέλουν ευρωπαϊκό μηχανισμό θέλουν να ξαναγυρίσουν σε μια ε, ξεπερασμένη διακυβερνητική προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, κατηγορώ το Συμβούλιο διότι μας ε, ε, φέρνει στα άκρα όπως ακούσαμε και από τους ομιλητές σήμερα. Είναι απαράδεκτο να γίνει επανεθνικοποίηση του εγχειρήματος Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ε, ζητεί να απαντήσει σύντομα. Παρακαλώ κύριε Μπότσκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μετά από την παρέμβαση του κυρίου Κοέλιο να τον ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε μαζί του, πολύ στενή συνεργασία. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κύριο Κοέλιο γιατί ήταν πραγματικά ουσιαστικός συμμέτοχος στις διαδικασίες λήψης απόφασης του Συμβουλίου. Παναλαμβάνω, το Συμβούλιο άκουσε τις διαφορετικές σας απόψεις, θα τις συζητήσουν εκ νέου στο Συμβούλιο και ελπίζω να μπορέσουμε επί τη βάση αυτών των θέσεων να προχωρήσουμε σε ένα επικοδομητικό διάλογο που θα διασφαλίσει την τεράστια προσπάθεια ενίσχυσης της διαχείρισης του Σέγγεν. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση